So. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Έχετε τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Όχι. Οπότε εγκρίνονται τα πρακτικά. Επόμενο σημείο είναι συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, οπότε δίνω σε τον λόγο στην κυρία Ντυραών για δύο λεπτά.